Good afternoon, colleagues. Um, we'd like to... Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Μπλίνκεβισιούτα και εγώ θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την κοινή συνάντηση των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΦΕΜ. Να σας ενημερώσω μόνο ε, τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ότι στις 5 θα παραταθεί η συνάντησή μας, αλλά θα πάμε σε άλλη αίθουσα, στην 4Q2. Θα φύγω λοιπόν κατά τις 5 παρατέταρτο, παρά 10 για να πάω στην άλλη αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν να γνωρίζετε ότι η συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα συνεχιστεί στην αίθουσα 4Q2 από τις 5 μέχρι τις 7. Ναι, ναι, μέχρι τις 7 θα συνεδριάσουμε. Να το ξέρουν αυτό οι συνάδελφοι της Επιτροπής Γυναικών, έτσι, αστιάκια κάνουμε. Okay, colleagues, um, so just... Λοιπόν, συνάδελφοι, Αυτά προς ενημέρωσή σας και καλώς ήλθατε σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΦΕΜ. Η συνεργασία των δύο επιτροπών μας ήταν πάντα εξαιρετική. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία για πολλά χαρτοφυλάκια, σε πάρα πολλά θέματα νομοθετικής και μη νομοθετικής ε, πρωτοβουλίας. Και τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολη για την πρόληψη και καταπολέμηση τη βίας κατά των γυναικών. Δημοσιεύτηκε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής συνάντησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να καταπολεμήσει την βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο συνεχίζονται και η Μαλτέζικη Προεδρία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και φυσικά το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει στη δουλειά αυτή με μια κοινή ενδιάμεση έκθεση. Στις 29 Νοεμβρίου του 2016 έγινε μια πρώτη κοινή συνάντηση για τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης και σήμερα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες στην ε, στο θέμα της καταπολέμησης της έμφυλης βίας για το διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Αυτά από την πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σχετικά με την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, κυρία Μπλίνκεβισιουτέ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράες. Αγαπητοί συνάδελφοι και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Γυναικών, Καλησπέρα σας, αγαπητοί εμπειρογνώμονες ε, που θα συμμετάσχετε στην ακρόαση. Καλώς ήλθατε όλοι στη σημερινή συνεδρίαση. Είναι η δεύτερη ακρόαση για ένα πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό ζήτημα. Την προσχώρηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η έμφυλη είναι στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής Γυναικών και Έχουμε ζητήσει πάνω από μία φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν σε αυτή τη σύμβαση. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ που επιτέλους δημοσιεύθηκε η πρόταση προσχώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπογραφεί και να ολοκληρωθεί η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση. Και οι δύο επιτροπές μας έχουν ένα μακρύ ιστορικό εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε αρχίσει δουλειά σε αυτό το θέμα πολύ καιρό πριν με την έκθεση της κυρίας Παρβανόβα η οποία παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει μέτρα κατά της έμφυλης βίας. Και, δίχως περαιτέρω καθυστερήσεις, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον, στην πρώτη προσκεκλημένη μας, την κυρία Σαχή Μπαγκαφαρόβα, η οποία είναι Γενική Εισηγήτρια για τη Βία κατά των Γυναικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Ορίστηκε Γενική Εισηγήτρια τον Απρίλιο του 2015 και κύριος ρόλος της είναι η ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Ευαισθητοποίηση και στο γενικό κοινό και ε, στα θεσμικά και μη θεσμικά όργανα και να προωθήσει την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης είναι πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ε, γυναίκες, τα παιδιά και την οικογένεια. Και επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής για γυναίκες, παιδιά και οικογένεια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαι εδώ, εκπροσωπώ την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κοινοβούλια να ενώσουν τι δυνάμει του τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώ για την καταπολέμηση τη βία σε βάρο των γυναικών και την πρόθεση των εργαλείων και μέσων που θα οδηγήσουν ε, στην ε, εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Φυσικά και χαιρετίζω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη Επίση, χαιρετίζω την απόφαση της Κομισιόν μέχρι το 2017 ε, να συνεχίσει προσπάθειες για την καταπολέμηση της βίας και να είναι και το έτος το 2017 φερωμένο στο σκοπό αυτό. Οι γυναίκες πλήττονται σε όλες τις χώρες από αυτό το φαινόμενο και όλοι μας, όλες μας έχουμε στον ευρύτερο ή στενότερο κύκλο ε, γνωρίσει θύματα ενδοκογενειακής βίας, έμφυλης βίας. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε και αν δεν το γνωρίζουμε δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα φύλου αν υπάρχει ένα μέρος του πλήσου που ζει μέσα σε φόβο και πανικό η ελευθερία από τη βία είναι προϋπόθεση για την ισότητα. Η καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών σημαίνει καταπολέμηση της ε, ανισότητας των φύλων. Η σημασία τη Κωνσταντινούπολη θεωρείται σταθμό στην προσπάθεια για την καταπολέμηση τη ενδοκογενειακή ευβία βία κατά των γυναικών. Είναι αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών ετών. Εμεί, ε, κυβερνήσει, εθνικοί βουλευτέ και των πολιτών, ε, εργαζόμαστε και στο μέτωπο τη ε, πρόληψη, Θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και μάλιστα τον Αύγουστο του 2014 πετύχαμε τον πρώτο μα στόχο όταν τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση ε, που θέλαμε να έχουμε. Γιατί η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση βελτιώνει την κατάσταση τη αντιμετώπισης του φαινομένου. Υπάρχουν πολλοί για του οποίου είναι τόσο σημαντικό αυτό το μέσο, αυτή η σύμβαση. Γιατί αναγνωρίζεται ότι είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακριτική μεταχείριση βία σε βάρο των γυναικών. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που περιλαμβάνει ορισμό του φύλου, ορίζει ε, τι αξιόπινε πράξει αυτέ, οι δεν περιλαμβάνονται ακόμη σε όλα τα εθνικά νομοθετικά πλαίσια, όπω είναι ο κολλητισμό γυναικείων, γεννητικών οργάνων, στόλ και τη βία, σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, βιασμό και εντό γάμου, ε, στήρωση, καταναγκαστική κτλ. κτλ. Έχουμε και μια επιτροπή στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου Ευρώπη. Προετοιμάζουμε ε, διάφορα ψηφίσματα κατά τη κακοποίηση, εξαλτική παρενόχληση, καταναγκαστικών γάμων. Ένα σημαντικό στοιχείο τη σύμβαση επίση είναι το γεγονό ότι ε, η παράδοση ή η τιμή, όπω λέγεται, δεν μπορεί να παρουσιάζεται πλέον ω αιτιολόγηση για την άσκηση βία και ε, αυτή την προσέγγιση την υποστήριξε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Επίση, η Σύμβαση αναφέρει κάποιες πρωτοβουλίε, εκπαίδευση επαγγελματιών, συλλογή δεδομένων, ε, επαρκή καταφύγια, γραμμές βοήθειας ε, Όλοι οι κρατικοί φορείς, όλε οι υπηρεσίε θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο τρόπο και αυτό σημαίνει ότι οι διάφοροι φορείς, ΜΚΟ, δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένοι στην δράση του. θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα συνεργασία. Ε, Στόχο τη σύμβαση είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκε, ε, η ασφάλεια των θυμάτων είναι στο επίκεντρο των μέτρων που λαμβάνονται. Πρόκειται για έναν σταθμό, για ένα ορόσημο. Θέτει σημαντικά ψηλά πρότυπα το τομέα τη προστασία, παροχή βοήθεια στα θύματα. Δίωξη των θητών. Συντονισμένε πολιτικέ. Μία από τι βασικέ προκλήσει τώρα σήμερα ποια είναι. Να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση για το πόσο κατεπήγον είναι αντιμετωπιστεί η βία σε βάρο των γυναικών. Τα κράτη θα πρέπει να δώσουν την απαιτούμενη υποστήριξη στα θύματα, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα τώρα να στραφώ στο συγκεκριμένο ρόλο των βουλευτών για την ε, διάδοση ε, των στόχων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Εγώ πιστεύω ότι κάθε βουλευτής μπορεί να αναλάβει το πρώτο δράση, όχι μόνο για την πρόθεση της Σύμβασης, αλλά και γενικά για την καταπολέμηση της βίας σε των σε εθνικό επίπεδο. Οι βουλευτές μπορούν να προωθήσουν την νομοθετική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υπογραφή και επικύρωση της Σύμβασης θα πρέπει να ζητήσουν τις κυβερνήσεις τους να οργανώσουν συζητήσεις, ε, να πάρουν πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και μεταξύ ΜΚΟ. και να προτείνουν και αναφορές, petitions για την υποστήριξη αυτής της σύμβασης συλλογή δεδομένων για τα φαινόμενα κατά βίας κατά των γυναικών. Ε, θα πρέπει να ζητήσουν επίσης χρηματοδότηση επαρκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι βουλευτές είναι ενεργοί ε, παράγοντες για την αλλαγή νοοτροπίας. Ε, γι' αυτό μπορούν να το πετύχουν αν υψώσουν το αναστημά του κατά τη βία αγορά των γυναικών, αν ασχίσουν πίεση και μέσα στα κόμματά τους για περισσότερη δράση με βάση τις ε, διατάξει της ε, σύμβασης, ε, οι βουλευτές συμμετέχουν άμεσα στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συνθήκης και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την υποβολή εκθέσεων των κρατικών φορέων, τις οποίες θα πρέπει να μελετούν, αλλά και ως ό,τι αφορά πληροφορίες που είναι τα κοινοβούλια. Διπλό ο ρόλο των βουλευτών. Σε εθνικό επίπεδο, τα κοινοβούλια μπορούν να παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνουν οι κρατικοί φορεί για την εφαρμογή τη συνθήκη. ευρωπαϊκό επίπεδο, Έχουμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, η οποία καλείται σε τακτά διαστήματα να κάνει τον απολογισμό τη εκτέλεση τη σύμβαση και μπορεί έτσι να αναφέρει τι ανησυχίε τη ό,τι αφορά πιθανέ αδυναμίε, ελλείψει ε, και για το πώ μπορούν συγκεκριμένε διατάξει τη συνθήκη να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό είναι ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο του ε, πολύ σημαντικού αυτού νομοθετήματο που ουσιαστικά είναι προ όφελο όλων. Οι αιρετοί δηλαδή άρχοντε να μπορούν να δίνουν τη συμβολή του ε, σε αυτό το πολύ σημαντικό συνθήκων για την παρακολούθηση δηλαδή της εφαρμογής της συνθήκης της σύμβασης. Ε, ως πολιτική συντονίστρια θέλω να μιλήσω για το κοινοβουλευτικό ε, δίκτυο Women Free From Violence. Αποτελείται το δίκτυό μας από βουλευτές που προέρχονται από 47 κράτη που είναι μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Είμαστε ε, στο, προσιλωμένοι στο στόχο της καταπολέμησης της ε, βίας βάση Είναι πολύ γνωστό το δίκτυο, δραστηριοποιείται με δηλώσει υψηλού επίπεδου σε εθνικά ε, κοινοβούλια είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, ένα εταίρο για το έργο τη Βουλή τη Ευρώπη. στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει την ενδοκογενειακή βία και τη των γυναικών. Τα δέκα χρόνια ε, πάνε από τότε που ιδρύθηκε το δίκτυο 2006. Έχει εξελιχθεί εκ τότε, έχει μεγάλη επίδραση με άλλου κοινοβουλευτικού φορεί και με διεθνεί οργανισμού όπω είναι η Κοινοβουλευτική Ένωση και το UN Women. Και βέβαια θέλουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με περισσότερε ανταλλαγέ σαν και αυτή μελλοντικά. Τα επόμενα χρόνια το δίκτυο θα συνεχίσει να αυξάνει την ορατότητα και τον αντίκτυπο του έργου τη συνέλευση στον τομέα τη καταπολέμηση τη βία σε βάρο των γυναικών. Θα οργανώσουμε εθνικά σεμινάρια, περιφερειακέ διασκέψει, τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν σε, κοινά, σε κοιν, μεικτέ Βασικός στόχος θα παραμείνει βέβαια προώθηση της υπογραφής επικύρωσης και εφαρμογή ε, της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Ε, το δίκτυο έχει να διαδραματίσει ένα ζωτικό ρόλο για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των βουλευτών για χώρες οι οποίες θα υποβληθούν σε παρακολούθηση. Θα πρέπει να τους δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία Έχουμε πρόσωπο του ΜΚΟ σήμερα στο πάνελ. Θα ήθελα να αναγνωρίσω το έργο των ΜΚΟ και να ευχαριστήσω τις ΜΚΟ για αυτό, γιατί εμείς ως βουλευτές βασιζόμαστε στην εμπειρία των ΜΚΟ για την εξέταση της ε, κύρωσης και εφαρμογή στη σήμανση στα Εθνικά Κοινοβούλια και τα μη, οι ΜΚΟ θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τα θύματα. Για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, θα πρέπει εμεί ω βουλευτέ να ασκήσουμε επιρροή, να μπορούν να έχουν την επαρκή χρηματοδότηση για προληπτικά μέτρα, για την παροχή βοήθεια και για τι ε, υπηρεσίε παροχή βοήθεια στα θύματα βία. Ολοκληρώνοντας κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι ως βουλευτές έχουμε μια μεγάλη δύναμη. Μπορούμε να επικοινωνούμε. Έχουμε χρόνο αγόρευση ε, στο ημικύκλιο και στα μέσα ενημέρωση. Αυτό το χρόνο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε μηνύματα, να πείσουμε το ακροατήριο ότι η βία σε βάρο των γυναικών είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Με τα λόγια μα μπορούμε να βοηθήσουμε τα θύματα ε, που δεν έχουν φωνή, να σπάσουμε τη σιωπή. Εμείς οι βουλευτές δεν θα πρέπει να μείνουμε βέβαια στα λόγια, αλλά να περάσουμε και στα έργα, να φέρουμε αλλαγές. Η προσχώρηση της Ένωσης στην Σύμβαση ήταν μια πρόκληση. Και μεγάλη ευκαιρία όμως ταυτόχρονα η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης πράγματι προωθεί ένα, ένα κοινωνικό όραμα. Ε, το όραμα μιας κοινωνίας που επιθυμούμε, όπου η βία σε βάση των γυναικών δεν θα είναι πλέον ούτε θα συγχωρείται ούτε και θα ελαχιστοποιεί τη σημασία της. Σας παρακαλώ και εσείς να χρησιμοποιήσετε όλο το βάρος που έχετε και να αποστηρίξετε τα θύματα, να ζητήσετε αλλαγή. Συγκεκριμένε αλλαγέ να ζητήσετε. Όπω παραδείγματο χάρη πρώτα απ' όλα επικύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε την Ελιζαμπέτ Μαρό Μπροντ. Είναι δικαστικός και Γενική Γραμματέα τη Διυπουργική Αντιπροσωπεία για την Προστασία των Γυναικών κατά τη Βία και την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων στη Γαλλία. Ο φορέα αυτό συλλέγει, αναλύει και δημοσιεύει πληροφορίε και δεδομένα στον χώρο τη βία κατά των γυναικών. Επίση, συμβάλλει στην αξιολόγηση των εθνικών και τοπικών μηχανισμών που λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο. Κυρία Μουαρόν Μπροντ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πρώτα απ' όλα να σα ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σα σε αυτήν την συζήτηση και συνεδρίαση που θα μας επιτρέψει, ελπίζω, να μοιραστούμε τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει για τα βήματα πρόοδου και τη συνεισφορά που πρόσφερε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι αλήθεια ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ε, της, του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών και της ενδογενειακής, η λεγόμενη δηλαδή της ε, Κωνσταντινούπολης, αποτέλεσε για τη Γαλλία ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που επιτρέπει να στηρίξουμε και να προχωρήσουμε έτσι την προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Να θυμίσω ότι η Γαλλία από πολλά χρόνια έχει θεωρήσει δημόσια πολιτική αυτή καθεαυτή την ε, πολιτική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Με την ενίσχυση του νομοθετικού μας οπλοστασίου και την ε, έγκριση τουλάχιστον πέντε τριετών σχεδίων και διυπουργικών σχεδίων και προγραμμάτων για το θέμα αυτό. Θα μιλήσω για την ενίσχυση του εθνικού μας οπλοστασίου που προϋπήρχε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δύο σημαντικοί νόμοι, θα αναφέρω τους πιο σημαντικούς, της Απριλίου 2006 για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στα πλαίσια του ζευγαριού, ε, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής των επιβαρυντικών στοιχείων για τις πράξεις βίας κατά του συζύγου και αυτό αφορούσε και τα ζεύγη που βρίσκονταν σε νόμιμη συμβίωση, όχι απλώς σε γάμο αυτό που ονομάζουμε στην Γαλλία ΠΑΞ. Και επίση του πρώην συζύγου. Αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία επίση διευρύνθηκαν περιλαμβάνοντα και άλλα στοιχεία πέρα από τι καθημερινές πράξεις βία, όπω ο φόνο, ο βιασμό και η σεξουαλική επίθεση. Ο νόμος αυτός είχε να κάνει και με την ε, απομάκρυνση του αυτούργου από την οικογενειακή αιστεία. Υπάρχει και ο νόμος της 10 Ιουλίου 2010, ο οποίος έχει να κάνει με τις πράξεις βίας κατά των γυναικών, τις πράξεις βίας εντός του ζεύγους και των πράξεων βίας κατά των παιδιών. Έτσι δημιουργήθηκε ένα εργαλείο προστασίας, πολύ, ιδιαίτερα πολύτιμο, που επιτρέπει στο δικαστή να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσει όποιον μέσα σε ένα ζεύγος μπορεί να είναι θέμα, θύμα ε, βίας. Ακόμη προβλέπεται και η πλήρης ε, αναστολή της γονικής κοκκιδαιμονίας για οποιονδήποτε είναι αυτουργός ή ύποπτος για την πράξη βίας κατά του προσώπου του άλλου γονέα. Και υπάρχει βεβαίως η πρόβλεψη και για το ποινικό αδίκημα της ψυχολογικής βίας, κάτι που το προβλέπει έτσι και η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ήθελα να πω ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πραγματικά είχε ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στην δημόσια πολιτική της Γαλλίας. Και αυτό θα ήθελα να το αναπτύξω σε τρεις άξονες ως θέμα, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, με την θέσπιση νέων θεσμικών φορέων, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ο δεύτερο άξονας είναι οι νόμοι που εγκρίναμε για να μεταφέρουμε στο δίκαιό μας τα πρότυπα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη για την προστασία των θυμάτων και την δίωξη των ε, δραστών. Τέλος, θα ολοκληρώσω με τον τρίτο άξονα για να σας εξηγήσω ότι πραγματικά σήμερα, χάρη στη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, γινόμαστε μάρτυρες μια πραγματική αναγνώριση που έχει ενταχθεί ε, πολύ, με πολύ γερά θεμέλια στο νομοθετικό τοπίο της Γαλλίας για την καταπολέμηση της βίας ειδικά κατά των γυναικών και το πεδίο ε, αντίδρασης ε, με πολύ συγκεκριμένου ορισμούς και πλαισίωση για αυτό το είδους βίας. Για τον πρώτο λοιπόν άξονα είναι οι θεσμικοί φορείς. Στι 3 Ιανουαρίου 2013, ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία ενέκρινε ένα ε, διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, για την ε, δημιουργία παρά του Υπουργείου που ασχολείται με τα θέματα των γυναικών, μια ε, διπουργική αντιπροσωπεία για την προστασία των γυναικών από τη βία και την καταπολέμηση τη εμπορία των ανθρώπων, η οποία ονομάζεται Μικρόφ. Και έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι διευθύντρια από τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Όπω το θυμήσατε κι εσεί, πρόεδρε, η Μικρόφ ασχολείται με τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των πληροφοριών και των δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών. Επίσης, ε, έχει ως έντολη στις αρμοδιότητές της να δημιουργήσει με τα Υπουργεία, την κοινωνία των πολιτών ένα ε, κατάλογο προτεραιοτήτων για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επιμένω στη διπουργική διάσταση της ΜΙΠΡΟΦ, της αντιπροσωπείας αυτής, η οποία είναι ένα, φανταστη... είναι ένα ε, αποφασιστικό πλεονέκτημα για να προαχθεί δράση ε, στον αγώνα της βίας κατά των γυναικών. το Υπουργείο για τη Δικαιοσύνη και τις Ελευθερίες και το άλλο για τις ε, γυναίκες είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά όλα τα Υπουργεία, όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, ε, το δικαστικό σύστημα, το σύστημα της δικαιοσύνης, το σύστημα υγείας και τους κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με την προστασία των θυμάτων. Οι αρμοδιότητα λοιπόν της Μικρόφ, της Μικρόφ μέσω του άρθρου 10 που προβλέπει ένα όργανο συντονισμού και 11 που προβλέπει τη συλλογή των δεδομένων είναι ξεκάθαρες. Αλλά υπάρχει και το άρθρο 15 λόγου χάρη που προβλέπει την κατάρτιση των επαγγελματιών. Από την δημιουργία της αντιπροσωπείας αυτή η Μικρόφ έχει αξιοποιήσει πολλά εργαλεία για την επαγγελματική κατάρτιση λόγου χάρη ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό ε, σύνολο ε, κοινών γνώσεων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, για όλους τους εργαζόμενους, για την, το εννοούμε με τη βία, την ενδοοικογενειακή για να δούμε πώς μπορεί να ε, υπάρχουν συνέπειες από την τραυματική εμπειρία πώς μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα τα θύματα και πώς μπορούμε καλύτερα να τα φροντίσουμε, να τους προσφέρουμε την ε, περίθαλψη που χρειάζονται στη συνέχεια. Τα εργαλεία που διαθέτουμε έχουν ε, δημιουργηθεί ανάλογα με την επαγγελματική κατεύθυνση των διαφόρων εργαζομένων. Δηλαδή, έχουμε ειδική κατάρτιση για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, για τους που εργάζονται στις ε, διοκτικές αρχές, ε, αστυνομικούς, χωροφύλακες, για τους δικαστικούς λειτουργούς, για τους κοινωνικούς λειτουργούς επίσης. Και Έχουμε και άλλα εργαλεία, ώστε πέρα των μορφών ενδοοικογενειακής βίας και άλλες μορφές βίας, όπως λόγου χάρη η σεξουαλική βία ο ακροτεριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων ή ο ε, καταναγκαστικός γάμο να προβλέπονται και αυτά. Και στο επίπεδο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση τη βία ε, κατά των γυναικών, έχουμε προβλέψει ένα πρόγραμμα εκπαίδευση ώστε να συγκεντρώνται σε κεντρικό επίπεδο όλε οι πληροφορίε, οι οποίε συστηματικά δημοσιεύονται στην ανάλογη εφημερίδα. Εφημερίδα τρίμηνιαία, η οποία δημοσιεύεται και στο, ε, στον ιστότοπο stopviolencefam.fr. Επίσης δημιουργήθηκε ο Φορέας για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2013 που αξιολογεί τις κρατικές πολιτικές ε, στο επίπεδο των ε, δικαιωμάτων των γυναικών με πέντε θεματικές ε, αρμοδιότητες. Πρώτα απ' όλα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών συγκεκριμένα με κρατικούς λειτουργούς δημοσίως δηλαδή υπαλλήλου και φορείς να δικτυώνονται μεταξύ του για να συζητήσουν τα θέματα αυτά και τη συνεργασία τη κοινωνία των πολιτών και των ε, αρμόδιων εμπειρογνωμόνων. Η δημιουργία αυτών των δύο φορέων ήταν πολύ σημαντική διότι όπω και εσείς θυμήσατε όχι μόνο χρειάζονται δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα για να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο, αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους επαγγελματίε και όλες οι κρατικές και δημόσιες πολιτικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές μόνο να αξιολογούνται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό. Αυτό ε, συμβαίνει με, την, με το Συμβούλιο για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Σε ό,τι αφορά την προστασία μας, ε, την νομοθετική, χάρη στα πρότυπα της Σύμβασης του Κωνσταντινούπολης, να θυμίσω την ε, το νόμο της 5ης 2013 που μιλά για την ε, βία, τις μορφές βίας και καθώς και για τον ακροτηριασμό των γυναικείων οργάνων ε, στις ανήλικες, στα ανήλικα κορίτσια. Έτσι θεωρείται ως ποινικό αδίκημα ακόμη και η επιβολή καταναγκαστικού γάμου, ακόμη και αν αυτό γίνει στο εξωτερικό και κάποια κοπέλα αναγκαστεί να φύγει από την επικράτεια τη Γαλλική Δημοκρατία. Προβλέπεται ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ. Επίση υπάρχει και ο νόμο τη 4ης 8-2015 για την ισότητα ανδρών και γυναικών που δίνει στο δικαστή τη ε, δυνατότητα να ε, προβλέψει ένα σεμινάριο για την ανάληψη ευθυνών στην περίπτωση που ε, υπάρχει μορφή βίας ή για την, αναστολή της γονικής κυδαιμονίας εφόσον ένα γονέα είναι ύποπτο, έχει διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει μορφέ βία κατά του παιδιού του και η ποινική και δικαστική διαμεσολάβηση στην περίπτωση μορφών βία στο πλαίσιο του ζεύγου στο άρθρο 8 τη ε, Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και που ουσιαστικά δεν είναι γενικότερο χαρακτήρα σε ένα σύστημα προστασία που ονομάζεται τηλεφωνικό αριθμό για σοβαρέ μορφέ βία. Σε περίπτωση που υπάρχουν μορφέ βία στην, ε, στο ζευγάρι και ε, ακόμη και διασμός και ο νόμος της 16ης Νοεμβρίου 2016 για διάφορε μορφές βία από του γονείς. Και ακόμη ένα νόμος το 2016 16, για την προστασία αλλοδαπών θυμάτων που μπορεί να έχουν ε, το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου ή του προσωρινού κατοίκου αλλά να είναι ε, σε ένωση νομική με κάποιον Γάλλο πολίτη. Τέλος, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προβλέπει την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των μορφών βίας κατά των γυναικών. Ως εκ τούτου την ανάγκη να προβλεφθεί μια ειδική πολιτική για τα θέματα αυτά. Η ιδιαιτερότητα αυτή βασίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα η βία κατά των γυναικών έχει να κάνει με την ισότητα ανδρών και γυναικών και πιο συγκεκριμένα οι μορφέ βία εντό του ζεύγου, οι σεξουαλικέ μορφέ βία, ο ακροτηριασμό των και γενετικών οργάνων και η εξανακαταστική γάμη έχουν να κάνουν με τι κοινωνικέ σχέσει και τη θέση των γυναικών σε σχέση με του άντρε. Καταλήγουμε στη διαπίστωση, διαπίστωση τη δυσανάλογη ε, θέση των γυναικών και των κοριτσιών που είναι εκτεθειμένε περισσότερο σε μορφέ βία, που δικαιολογεί αυτό και την ιδιαιτερότητα αυτών των μορφών βία. Οι γυναίκε είναι το 85% θυμάτων ενδοικογενειακή βία ή ε, θύματα εντό του ζεύγου επίσης ε, σε πολύ ψηλά ποσοστά. Κάτω των 15 ετών μορφές βίας διαπιστώνονται από την αστυνομία και του, τις δικτικές αρχές κατά των γυναικών. Επίσης να πω ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μας επιτρέπει να μελετήσουμε στα πλαίσια της καθημερινής μας δουλειάς τα θέματα αυτά. Λόγου χάρη να αναφέρω την ε, συνειδητοποίηση αυξανόμενη συνειδητοποίηση στη Γαλλία το πόσο ε, οι μορφέ βία εντό του ζεύγου έχουν αντίκτυπο και στα παιδιά. Το πέμπτο μα πρόγραμμα που εγκρίθηκε στι 5 Νοεμβρίου πέρσι και το πρώτο πρόγραμμα δράση για τι μορφέ βία κατά των παιδιών λαμβάνουν υπόψη και τα δύο αυτόν τον τόσο σημαντικό αντίκτυπο που τονίστηκε και από την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ιδού, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Απλώ να σα πω ότι η τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2014 Ήταν πολύ σημαντική γιατί μας επιτρέπει να ε, δούμε σε μακρινό ορίζοντα ακριβώς τον, ε, την πολιτική μας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις πραγματικές ανάγκες της ισότητα ανδρών και γυναικών. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπρο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Γκουνχάιμερ. Ο καθηγητή Χάιμερ είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Γνώσης για τη Βία των Ανδρών κατά των Γυναικών ε, του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία. Είναι ένα κέντρο που διευθύνει από κοινού το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλα και εκτός από θέματα βίας κατά των γυναικών ασχολείται με μεθόδους πρόληψης ε, της έμφυλης βίας. Καθηγητά Χάιμερ, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Καθηγήτρια Χάιμερ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που κάνατε στο κέντρο μας να βρεθούμε στην ακρόαση αυτή. Καταρχάς, να σας πω ότι βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο της ουψάλα και η εντολή μας προέρχεται από την κυβέρνηση της Σουηδίας. Συλλέγουμε γνώση, παρέχουμε κατάρτιση και διεξάγουμε ερευνητικό έργο, κατάρτιση για φοιτητές και επαγγελματίες, ε, δίνουμε στήριξη σε διάφορες κυβερνικές οργανώσεις και τέλος τις ίδιες τις γυναίκες πέφτουν θύματα έμφυλης βίας. Τώρα, να σας πω δύο λόγια για τη δομή μας. Είμαστε το πρώτο τέτοιο κέντρο στην Σουηδία. Δημιουργηθήκαμε το 1994. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Είναι το μεγαλύτερο στη Σουηδία. Και επίσης παρέχουμε κατάρτιση, διεξάγουμε έρευνες και ανάλυση για θέματα εμφυλη. Οι μελέτες μας δημοσιεύονται κιόλα και κέντρο των ερευνών μας είναι μία μελέτη για το έβρο της έμφυλης βίας στην Σουηδία. Ασχολούμαστε με την σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική βία που υφίστανται γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και Είμαστε επίσης σε επικοινωνία με γυναίκες που έχουν υποστεί βία και την έχουν ξεπεράσει. Τώρα, η έκθεση στη σεξουαλική βία. Ε, κατά τη διάρκεια της ζωής της, ε, μία ε, γυναίκα υφίσταται σεξουαλική βία. Πάνω, 25% των γυναικών είναι το ποσοστό που υφίσταται βία. Τώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σουηδίας ανέθεσε στο κέντρο μας να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα στήριξης και διαχείρισης των θυμάτων της έμφυλης βίας, να παρέχει ιατρική και ψυχολογική ε, βοήθεια και να καθορίσει το ρόλο των υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια μιας ε, δικαστικής διαδικασίας έμφυλης βίας. Μετά. Το κέντρο μας δημιούργησε ένα ε, kit ταυτοποίησης της σεξουαλικής βίας. Έχουμε ένα σύνολο εργαλείων για τον εντοπισμό ε, περιπτώσεων σεξουαλικής βίας, το οποίο χρησιμοποιούν οι γιατροί στις εξετάσεις τους. Ε, τους παρέχουμε κατάρτιση για το τι πρέπει να κάνουν και πώς. Αυτό αυτή η κατάρτιση παρέχεται στους επαγγελματίε υγείας τόσο για τις γυναίκες θύματα όσο και για τους άνδρες θύματα και ε, είναι διαθέσιμο σε όλη την επικράτεια της Ουδίας από τον Ιανουάριο του 2011. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, οι επαγγελματίες υγείας ε, και είναι αρκετά εύχριστο. Μετά, όπως σας είπα, υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το hotline Κβίνο Λίνιεν στα Σουηδικά λέγεται. Το κέντρο αυτό το διαχειρίζεται η κλινική μας. Έδρα έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλα. Άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2007 και λαμβάνει πάνω από 31.000 κλήσεις ετησίως. Και φανταστείτε το μέγεθος, ε, να σας πω μόνο ότι ο πληθυσμός της Σουηδίας είναι 10 εκατομμύρια. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Από επαγγελματίες οι κλήσεις είναι δωρεάν και δεν εμφανίζονται στην αναλυτική, στον αναλυτικό λογαριασμό κλήσεων ε, του σπιτιού και παρέχουμε πληροφορίες στις γυναίκες για διάφορα καταφύγια που μπορούν να πάνε, κοινωνικές υπηρεσίες, ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ. Υπάρχει πρόσβαση των γυναικών σε διερμηνείς, μπορούν να μιλήσουν πολλές γλώσσες, υπάρχει ιστοσελίδα και ιστότοπος του κέντρου μας και οι πληροφορίες του κέντρου είναι διαθέσιμες σε 27 διαφορετικές γλώσσες. Ξεπερνάμε δηλαδή τι απαιτήσει τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Λαμβάνουμε περίπου 85 κλήσεις την ημέρα. Όπω βλέπετε και στη διαφάνεια, οι 72 από τι 85 είναι από γυναίκε που πέφτουν θύματα βία και οι 10 από ε, την οικογένεια ή του φίλου των ε, θυμάτων. Και οι 3 από τι 85 κλήσεις από επαγγελματίε που ζητούν περισσότερε πληροφορίε. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοθεί ένα τέλος στην ε, βία κατά των γυναικών. Το κέντρο μας, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, νομίζω πως ε, είναι αναγκαίο για να δοθεί λοιπόν ένα τέλος στη βία των γυναικών. Επίσης, δίωξη. Η βία κατά των γυναικών είναι ποινικό αδίκημα, είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Χρειάζεται επομένως ε, να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση έτσι ώστε να αυξηθούν οι διώξεις και ε, οι περιπτώσεις ε, προσφυγής στα δικαστήρια, να αυξηθούν οι καταδίκες επίσης ε, των φυτών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης τα θύματα να λαμβάνουν σωστή φροντίδα, περίθαλψη, ενημέρωση. Γι' αυτό διοργανώνουμε διάφορα πανεπιστημιακά μαθήματα για επαγγελματίε αλλά και για φοιτητέ ε, παρέχουμε εκπαίδευση, έχουμε διάφορα προγράμματα e-learning, ηλεκτρονικής μάθησης, ε, για τα οποία θα σας ενημερώσω σε λίγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Άννα και Έγκστρομ, τη συναδελφό μου, για να σας ενημερώσω σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η ένα αποτέλεσμα της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στην Σουηδία είναι ότι μας έχει αυξηθεί η ζήτηση για εκπαίδευση από επαγγελματίε ε, υγείας. Γι' αυτό λοιπόν το κέντρο μας συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας της Σουηδίας και τα επιμέρους ε, συμβούλια στις διάφορες περιφέρειες για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης ε, και ενημέρωσης για τη βία κατά των γυναικών. Είναι μια διαδραστική πλατφόρμα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν. Είναι δωρεάν η εκπαίδευση και πρόσβαση μπορούν να έχουν όσοι το επιθυμούν. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να γίνουν είτε ατομικά είτε σε group, έτσι ώστε να συζητηθούν μαζί με τους ε, συναδέλφους συμμετέχοντες σε διάφορα θέματα έμφυλης βίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Το σεμινάριο διαρκεί περίπου δύο ώρες. Είναι μια πολύ σύγχρονη μέθοδος ε, εκπαίδευσης. Υπάρχουν διάφορες συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, με επαγγελματίε και βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Επίσης, παρέχεται ενημέρωση για την νομοθεσία στη Σουηδία, για τις ε, συνέπειες τόσο τις νομικές όσο και στην υγεία και από τότε που άρχισαν αυτά τα online μαθήματα, υπήρξαν 8.500 εγγραφές, 172 ομάδες και τα μαθήματα αυτά έχουν τη δομή ενός ιστοτόπου. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, οι χρήστε είναι κατά το ίμιση άτομα που εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες και 16% ε, άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας. Οι υπόλοιποι είναι ε, υπάλληλοι τη αστυνομίας, ε, εισαγγελεί, δάσκαλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τα online μαθήματα έχουν μεγάλη επιτυχία, έχουν καταφέρει να αυξήσουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση ε, του κοινού στη Σουηδία και νομίζω πως η ευκολία χρήσης ε, οφείλεται, μάλλον και νομίζω πως οφείλουν την επιτυχία τους στην ευκολία χρήσης. Σας ευχαριστώ. Ε, ολοκληρώσατε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και τις δυο. Επόμενη είναι Μαρία Μιγέλ Σιέρα, που είναι διευθύντρια της Λαβάντε Φάμα, μια ένεση που ασκείται στο Βέλγιο Βρυξέλλες για την κοινωνική ένταξη και είναι και η πυρογνώμων του Βελγίου στο παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ και χρόνια η βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών είναι στο επίκεντρο του έργου του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών που έχει θεσπίσει εδώ και 20 χρόνια ένα παρατηρητήριο για τα φαινόμενα βία σε βάρος των γυναικών, με εμπειρογνώμονε, επαγγελματίε των κλάδων σε διάφορα κρατημέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά τα φαινόμενα βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τη συχνότητα αυτών. Είμαι διευθύντρια ενός ιδρύματος για τις μετανάστριες και η εμπειρογνώμων του Βελγίου ε, στο παρατηρητή. Θέλω λοιπόν και εγώ να πω πόσο σημαντικό είναι το εργαλείο αυτό της σύμβασης της ε, που τέθηκε ισχύει την 1η Ιουλίου του 2016 ε, στο Βέλγιο και ήδη βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου. Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Βελγίου είναι ότι διαρθρώνεται εξ ολοκλήρου με βάση τη δομή της ε, Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, με στρατηγικούς τομείς, που ουσιαστικά είναι οι ίδιοι ε, ένας μετά τον άλλον ε, με τους στόχους της σύμβασης της δεν θα για τα 135 μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2019 απλά θα ήθελα να περιοριστώ σε μια πτυχή που δεν έχει ληφθεί υπόψη ε, επαρκώς μέχρι σήμερα από τις βελτικές αρχές και μιλώ για τη σεξουαλική βία. Τι μας επιτρέπει ήδη η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να λάβουμε καλύτερα υπόψη τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας με την ανάπτυξη κέντρων για την υποδοχή των ε, θυμάτων. Έχουμε τρία πιλωτικά σχέδια στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Οι μερίδες μελέτης για τους αστυνομικούς, για τη σεξουαλική βία, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης διαχείρισης κινδύνων, ε, μια νέα ιστοσελίδα και καμπάνιες ευαισθητοποίησης μεγάλης κλίμακας. Και μιλάω για ένα μόνο θέμα, για να σας δείξω ότι με λίγη προσπάθεια μπορούμε, όπως ζητείτε στην σύμβαση, να αντιμετωπίσουμε με διαρθρωτικό, πολυεπίπεδο και διακλαδικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Από τότε που τέθηκε ισχύ η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, συνέβησαν σημαντικά πράγματα με την κινητοποίηση και όλων των ΜΚΟ. Καταφέραμε να διευρύνουμε, βελτιώσουμε τις δομές φιλοξενίας γυναικών που δεν είναι παρκισακόμη, ακόμη. Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε και θα ζητήσουμε περισσότερες θέσεις. Θέλουμε να υπάρχουν περισσότερες θέσεις και κάλυψη κάθε μέρα επί 24 ώρου βάσεως. Αυτό που είναι ήδη ενδιαφέρον είναι ότι η σύμβαση αυτή επέτρεψε σε μια δυναμική να αναπτυχθεί. Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της σύμβασης πρέπει να δημιουργηθούν κοινοπραξίες να υπάρξει συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων. Το βλέπουμε κάθε μέρα επί τόπου. Υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για το θέμα της βίας. Γίνεται λόγος για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει ακριβώς περί τίνο πρόκειται, αλλά σχετίζουν τη βία με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Και μιλώ για τη βία σε βάρος γυναικών κοριτσιών βέβαια. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Για να συνεχίσουμε να προκαλούμε το ενδιαφέρον και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Πανέρχομαι στο ευρωπαϊκό όμω επίπεδο γιατί εκπροσωπώ και το λόμπι των ε, γυναικών. 2017 είναι το έτος δράσης για την καταπολέμηση ασφάλειας των γυναικών. Η κυρία Γιούροβα, ε, επίτροπος, το πρότεινε. Και πρότεινε και την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Εμείς είμαστε πολύ ευγνώμονες γι' αυτό. Όλες οι δράσεις ε, που μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητες για την εκρίζωση της βίας σε των γυναικών. Η βία σε βάρο των γυναικών είναι η πιο συχνή παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συχνότητα δείχνουν ότι οι πατριαρχικές αξίες ε, και ο φαλοκρατισμός εξακολουθούν να είναι φαινόμενα πολύ δεδομένα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ευεξία, τον επαγγελματικό βίο, γιατί όλα αυτά είναι εμπόδιο για την ε, οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη συμμετοχή τους ε, στα κοινωνικά και τα δημόσια πολιτικά δρόμενα και ούτω καθεξής. Οι γυναίκες στα κορίτσια ε, πέφτουν θύμα βίας, στο ζευγάρι, στο δρόμο, στη δουλειά, στο διαδίκτυο. Να σας δώσω κάποια στοιχεία μόνο στην Ευρώπη. 50 γυναίκες την εβδομάδα πεθαίνουν από ενδοοικογενειακή βία. Στα χέρια αντρών, 35% τουλάχιστον έζησαν μια εμπειρία ε, φυσικής, σωματικής, ψυχολογικής βίας από την ηλικία των 15 και ένας στους 5 θεωρούν ότι τα θύματα φταίνε για τη βία ή ότι υπερβάλλουν, τα φουσκώνουν τα γεγονότα. 2,28 δισεκατομμύρια, το 2% του ΑΕΠ είναι το κόστος λόγω αυτών των ε, φαινομένων. Είναι ε, τραγικά αυτά τα νούμερα. Συνεχίζει όμως το φαινόμενο να θεωρείται τετριμένο. Δεν θεωρείται πολιτική προτεραιότητα. Υποβαθμίζεται. Τα τελευταία χρόνια τα μέτρα λιτότητας ε, οδήγησαν σε μείωση στον προϋπολογισμό στήριξης των θυμάτων και προληπτικών μέτρων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βία και η αποτυχία της κυβέρνησης να την αποφύγει είναι κάτι πολύ αρνητικό για τις γυναίκες και τις ε, κοπέλες. Το πολιτικό νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές σήμερα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ε, που θέτει το πρόβλημα αυτό. Οι ποινικοί κώδικε δεν ε, θεωρούν αξιόπινε πράξει όλε τι μορφέ βία των γυναικών. Υπάρχουν δε ειδικοί νόμοι που δεν, είναι πάντοτε, δεν συνοδεύονται πάντοτε από τα επαρκή μέτρα ειδικές υπηρεσίες, ε, για τις, ε, τα, τα καταφύγια, δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και συχνά τα διαχειρίζονται μη και όπου δεν έχουν ε, μόνιμη χρηματοδότηση. Οι επαγγελματίε που είναι σε άμεση επαφή με τα θύματα, κοινωνικοιατρικέ υπηρεσίε, αστυνομία, δικαστικό σώμα, δεν έχουν τη σωστή εκπαίδευση πολύ συχνά. Και πολλές φορές η αντιμετώπιση οδηγεί σε θυματοποίηση, δευτερογενή θυματοποίηση. Επίσης, τα διαρθρωτικά αίτια δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικο-οικονομικό ρόλος που ε, αποδίδεται σε άνδρες και γυναίκες. Έχουμε πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, ιδίως λόγω καταγωγή, ηλικία, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητα, ε, αν είναι μετανάστε ή όχι, θρησκεία και όλα αυτά. Δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώ. Πολλέ γυναίκες επειδή φοβούνται μην τι απελάσουν, ε, δεν ζητούν την προστασία τους. Και επίση υπάρχουν πάρα πολύ λίγα καταφύγια για μετανάστριες ή πρόσφυγε. Πόσο μάλλον για αυτέ που δεν έχουν καν χαρτιά. Τέλος οι γυναίκες, τα κορίτσια στην Ένωση δεν έχουν ισότιμη προστασία σε βάρος της, ε, μάλλον ε, από τη βία λόγω του ότι δεν υπάρχει ε, νομιογενείς πολιτικές και μέτρα στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική, αλλά δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο για την μετατόπιση της βίας σε βάρος των γυναικών. Η πραγματική ισότητα μεταξύ των και γυναικών θα μείνει ένα δράμα όσο δελείται το πρόβλημα της βίας σε βάρος γυναικών κοριτσιών με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι δεσμευτική. Έχει ολιστική, πολυεπίπεδη, διακλαδική προσέγγιση. Τονίζει λοιπόν την ανάγκη εταιρικών σχέσεων και καλύπτει τα κενά ε, στις εθνικές ε, προσπάθειες. Και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ε, στηρίζεται από 25 δίκτυα και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετεπιτάσεως να προσχωρήσει στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Έχουμε πάνω από 60.000 υπογραφές πολιτών υπέρ της προσχώρησης ως το δυνατόν ευρύτερης προσχώρησης Ένωσης στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Έτσι η διεθνή κοινότητα θα λάβει ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε προσιλωμένοι στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συλλογή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Θέλουμε επίσης να υπάρξουν προ, και πιο αποτελεσματικέ προληπτικές πολιτικές, να εμβαθύνουν, να βελτιώσουμε την προστασία των θυμάτων. Το λέει και οδηγία για τα θύματα. Για να έχουμε καλύτερο συντονισμό των πολιτικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά και για να διατεθούν οι απαρικοί σπόροι σε μόνιμη βάση. Πρέπει να σκεφτούν περαιτέρω πιέσει πολιτικέ στα κράτη-μέλη για να επικυρώσουν τη σύμβαση να υπάρξει καλύτερη δικαστική συνεργασία. Όπως ισχύει για το εμπόριο ανθρώπων. Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν κάνει μια κοινή διακήρυξη το Φεβρουάριο στη Μάλτα για μηδενική ανοχή στα φαινόμενα βία σε βάρος γυναικών κοριτσιών και αυτό περιμένουμε να γίνει πράξη και κατεπηγόντως. Προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μιγγέλ Σιέρα και τώρα να δώσω το λόγο στην στο ε, ε, τελευταία μέλη του πάνελ, δηλαδή τις δύο συνεισηγήτριες, είναι δύο, η κυρία Ρεβονταλόν Μπονφουά, και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Πρώτη, η κυρία Ριβονταλόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη κυρία Μπίλτ, η οποία δεν θα αργήσει, αλλά έχει ένα πρόβλημα με την πτήση τη. Οπότε συγχωρήστε την, ε, δεν φταίει εκείνη. Θα έρθει μόλι μπορέσει. Καταρχάς να ευχαριστήσω τις συμμετέχουσες στο πάνελ, οι οποίες ε, και έδεχτηκαν την πρόσκλησή μας και αγωνίζονται για την καταπολέμηση της φύσης κατά των γυναικών. Είναι μεγάλη μου χαρά και είμαι περήφανη που είμαι μαζί σας σήμερα και που βρίσκονται εδώ αυτές ε, οι εμπειρογνώμονες ε, που συμμετέχουν στην προσπάθεια να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Σύμβαση του Κωνσταντινούπολη. Χρειάζεται κοινή δουλειά των δύο επιτροπών μα για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε αναλάβει, δηλαδή να ε, ξαγλύψουμε την βία κατά των γυναικών, όποια μορφή βία και αν είναι αυτή, και σε οποιαδήποτε σφαίρα του δημόσιου του ιδιωτικού βίου. Το 2017 ο αγώνα αυτό είναι ακόμη αναγκαίο. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τη έρευνα του Παρατηρητηρίου για τα του δικαιώματα στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο αγώνα αυτό να συνεχιστεί. Ένα τρίτο των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική σεξουαλική βία στη ζωή του. Μία στι 20 γυναίκε έχει βιαστεί από τα 15 τη. Οι μισέ γυναίκε τη Ευρωπαϊκή ε, ε, ή σημεία και χώρους και ε, χώρου από φόβο μήπω δεχτούν σεξουαλική ήσωματική επίθεση. Αυτή η σημεια και χωρου απο φοβο μηπω δεχτουν σεξουαλικη άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για μια κοινωνία όπου ο μισό πληθυσμός έχει ένα μόνιμο κίνδυνο να υποστεί βία, να γίνει θύμα. Θα πρέπει ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του. Ο καθένα θα πρέπει να αισθάνεται τον αφορά το θέμα, όχι μόνο οι γυναίκε και τα κορίτσια. Είναι ύψη τη σημασία και οι άντρε και τα αγόρια να λάβουν γνώση του φαινομένου, αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα για τον ρόλο και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Ορισμένοι θεωρούν ότι η ε, ο εκφοβισμό μια γυναίκα, η επίθεση σωματική ή ψυχολογική δεν είναι μορφή βία. Κάποιοι θεωρούν ότι του αξίζει ατιμορρησία. Άλλοι δηλώνουν ότι οι σεξουαλικέ σχέσει χωρί τη συγκατάθεση τη γυναίκα μπορούν να δικαιολογηθούν. Αυτέ οι συμπεριφορέ είναι απαράδεκτε. Πολλέ φορέ τα θύματα δεν καταγγέλουν στην αστυνομία τη βία που έχουν υποστεί διότι φοβούνται τα αντίπεινα ή την ε, αντίδραση. Έτσι, οι φορείς δεν έχουν ανησυχήσει και έχουν καθυστερήσει να προβλέψουν ως ποινικό αδίκημα ή ως τη βία κατά των γυναικών. Θα έπρεπε όμω να ντρέπονται και να τιμωρούνται οι δράστε και οι αυτούργοι. Να θυμίσουμε ότι οι γυναίκε βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών διακριτικών μεταχειρήσεων. Αυτέ που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη βία είναι αυτέ που βρίσκονται σε θέση επισφαλή, ευάλωτη λόγω των σεξουαλικών του προσανατολισμών, τη ταυτότητα φύλου, τη ηλικία του, τη αναπηρία του, τη καταγωγή του. Ή αν είναι πρόσφυγε, μετανάστηδε ή ε, ετούντε άσυλο. Ετούσε μάλλον άσυλο. Θα πρέπει όλε ε, οι γυναίκε και τα κορίτσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατευθούν. Ε, μιλάμε από την αρχή του απογεύματο για τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Είναι το πρώτο εργαλείο που διαθέτουμε, που είναι διεθνέ και νομικώ δεσμευτικό για το θέμα. Ε, η σύμβαση αυτή δράζει πολλά επίπεδα, όπω την πρόληψη, την καταπολέμηση των, των μορφών διακριτική μεταχείριση, των ποινικών μέτρων, τη προστασία και τη στήριξη των θυμάτων, τη ειδική προστασία που προβλέπεται για τα παιδιά, αλλά και στου πρόσφυγε και τι αιτούσε άσυλου. οι ε, μορφές βίας κατά των γυναικών πρέπει να προβλέπονται, αλλά και οι πρόληψη, ε, αλλά ε, η καταπολέμηση όλων των μορφών είναι σημαντική. Η προστασία των θυμάτων, η δίωξη των αυτούργων και δραστών. Όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται μετά. Ε, γι' αυτό χρειάζεται η κύρωση τη σύμβαση για να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Η έκθεσή μα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει και να, προσυπογράψει την, να προσχωρήσει τη σύμβαση αυτό το δυνατόν συντομότερα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιφυλάξει ε, σε κανένα από τα κράτη-μέλη, διότι είναι πολλέ οι αρμοδιότητε τη Ένωση στο συγκεκριμένο τομέα. Το δίκαιο τη Ένωση δεν απαλλάσσει τα κράτη-μέλη από τι ευθύνε του. Ε, όσοι έχουν συνυπογράψει, μόνο 14 έχουν κυρώσει τη σύμβαση ω τώρα, να το θυμίσω, και είναι τελείω ανεπαρκέ. Όσοι έχουν λοιπόν συνυπογράψει πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Πρέπει μαζί να δημιουργήσουμε ένα συνεπέ νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να προστατεύσουμε όλε τι γυναίκε και τα κορίτσια όποιο και αν είναι ο τόπο διαμονή του στην Ευρώπη. Οι αντιδραστικέ ε, τοποθετήσει ορισμένων κατών μελών κατά των γυναικών ε, δεν δικαιολογούνται. Οι γυναίκε δεν είναι προστατευμένε έναντι τη βία ε, και δεν μπορούν να προστατεύονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα που κατοικούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια αναντήρητη συγκριτική αξία, ιδίω για τη σύγκριση των δεδομένων των μορφών βία στα θέματα της έμφυλης βίας, διότι μας λείπουν τα δεδομένα σε αυτόν τον τομέα. Η μάστιγα αυτή έχει πάρει πολλές, πολύ μεγάλες διαστάσεις. 30% των γυναικών στη Γαλλία λόγου χάρη ε, χρειάζονται και ιατρική περίθαλψη, αλλά δεν τα ζητούν πάντοτε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει απαραίτητη εκπαίδευση όσων εργάζονται στο κοινωνικό τομέα, ώστε να προστατεύουν και να περιθάλπουν ανάλογω τα θύματα. Πρέπει η κουλτούρα όλη τη Ευρώπη να αλλάξει, ώστε η απόκρισή μα να είναι εύστοχη, σκόπιμη και αποτελεσματική. Μόλι κυρωθεί η σύμβαση, δεν θα έχει λήξει ο αγώνα μα. Αντιθέτω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση και την πλήρη αφοσίωση όλων των απαραίτητων εργαλείων στην επίτευξη των στόχων μας. Πρέπει να προβλέψουμε απαραίτητα και ε, κατάλληλα μέσα, ώστε όλα αυτά τα μέτρα να πάρουν ένα και και να υπάρξει απαραίτητη πολιτική δράση. Είμαστε πεπισμένοι ότι μια οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση των μορφών βίας κατά των γυναικών θα είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να το προβλέψουμε. Η οδηγία αυτή θα δώσει κοινού ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα αδικήματα που διαπράττονται κατά των γυναικών, ώστε να ενισχυθεί η υλοποίηση τη σύμβαση και το πλαισιό και να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα μέτρα ή διατάξει που αφορούν τι αρμοδιότητε τη Ένωση. Εδώ κάνω, απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο που είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά. Έχει φτάσει η στιγμή, δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο για να γίνει κάτι. Το αναφέρει και η επιστολή μα του μηνό Φεβρουαρίου. Θα ολοκληρώσω επιμένοντα το εξή σημείο. Η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμφωση Κωνσταντινούπολη θα ε, ενισχύσει την καταπολέμηση τη βία και την ε, καθιέρωση τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπω προβλέπουν οι συνθήκε λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Δεν έγινε νοήματο αυτή η επιταγή. Είναι φιλόδοξη η στόχη που έχουμε θέσει, αλλά υπάρχει πολλή δρόμο που πρέπει να γίνει ακόμα. Ε, η έκθεσή μα δείχνει ε, την πολιτική δέσμευση του Κοινοβουλίου ε, να προστατεύσει τους μισούς πολίτες της Ένωσης στην ουσία. Ε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης προφανώς για τις προσπάθειε τους και την αφοσίωσή τους στον σκοπό αυτό και να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ με την ελπίδα και την τόλμη που έχουμε όλοι για να φτάσουμε στο τέρμα της διαδικασίας της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Um, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κριστίν. Προτείνω τώρα να ακούσουμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ όταν καταφέρει να φτάσει και στο μεταξύ να ακούσουμε τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στα δύο λεπτά και πρώτη έχει το λόγο η Μαλίν Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, τους εμπειρογνώμονες, όσους μίλησαν και τα ε, μέλη τη επιτροπή, τι εισηγήτριες και την κυρία Κορατσαμπίλη όταν αυτή έρθει για τη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Εμεί είμαστε υπέρ τη προσχώρηση τη σύμβαση Κωνσταντινούπολη, διότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ε, και με αφορμή αυτό σκεφτόμουν όλους ε, εκείνους που προσπάθησαν να κάνουν την ισότητα πραγματικότητα. Οι γυναίκες, οι, οι φεμινίστριες, εργαζόμαστε πολλά χρόνια γι' αυτό, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και ε, το ανέφεραν και πολλοί ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία συνεχίζει να αποδέχεται τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ε, πολλές φορές μας αρέσει να αναφερόμαστε στη βία, σε άλλους, άλλες κουλτούρες, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκατοντάδες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα εξαιτία της ε, έμφυλης βίας και πολύ σπάνια ε, υπάρχουν καταδίκες και οι καταδίκες αυτές δεν έχουν τις ποινές που θα έπρεπε. Και ε, νομίζω πως θα μιλάμε χωρίς να κάνουμε τίποτα αν συνεχίζουμε να μην αναλαμβάνουμε δράση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναλάβουμε δράση, να ανασκουμποθούμε έτσι ώστε να προσχωρήσουμε στην Σύμβαση Κωνσταντινούπολη και οι γυναίκε να απολαμβάνουν ισότητε και προστασίε όπω ε, του ε, αξίζει. Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά βέβαια. Έχουμε κάνει προπαρασκευαστικέ εργασίε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε οι ε, δράστε να διώκονται ποινικά και τα θύματα να προστατεύονται. Γι' αυτό πρέπει, πιστεύω, σε εθνικό επίπεδο να συλλέξουμε όλα τα, όλες τις καλύτερες βέλτιστες πρακτικές και υπάρχουν αρκετά ε, πολλά τέτοια καλά παραδείγματα στην Ισπανία, ας πούμε, και αλλού. Γιατί πραγματικά πρέπει να ε, βρούμε τις καλύτερες πρακτικές. Αυτό μας ζητάνε και περιμένουν από εμά οι γυναίκες και τα κορίτσια ως ε, νομοθέτες. Και όπω ε, είπατε, το θέμα δεν είναι μόνο η προσχώρηση στη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό είναι εύκολο, μπορούμε να, να το κάνουμε χωρί να αλλάξουν τα πράγματα. Χρειάζεται στρατηγική που θα εφαρμοστεί κατά τη ε, βία ε, κατά των γυναικών και των κοριτσιών των ΛΟΑΔ. Θέλουμε όμως πολλά περισσότερα. Νομοθεσία, όχι μόνο στρατηγική. Γι' αυτό λοιπόν θα ευχαριστήσω όλους εσάς για αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαρσία Πέρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες ε, που έλαβαν το λόγο στο πλαίσιο αυτής της ακράσης, ε, διότι αυτά που μας είπαν κυρίως ε, μας κάνουν να αντιληφθούμε πώς αποκρισταλώνονται αυτές οι ενεργές πολιτικές για την καταπολέμηση εμφυλής στα διάφορα κράτη-μέλη με τις διάφορες πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά υπόψη μας το πόσο ε, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ε, πληροφορίες που παίρνουμε εδώ για να υιοθετήσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές παίρνοντας το καλύτερο από τις πρωτοβουλίες και από την νομοθεσία των κρατών για να τα καταπολεμήσουμε την κοινωνική αυτή Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι ένα θεμελιώδη ζήτημα. Ουσιαστικά είναι η καταπολέμηση της φαλοκρατικής τρομοκρατίας. Γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους στα χέρια του συντρόφου τους, ε, του άντρα τους. Μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες ε, και επειδή δεν είναι η, κοινότητα, η κοινωνία στην οποία ζούμε δίκαιη και ίση, κάποιο ε, τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη ουσία σε σχέση με το άλλο τμήμα. Αυτό ε, είναι που ε, οδηγεί σε αυτή τη βία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις πολιτικές, αυτό είναι απαραίτητο, είναι επίγον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Όπως είπε όμως και συντρόφισσα η συγγήτρια, από το Κοινοβουλίο. Αυτό δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα, αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη να απεκδεθούν των δικών τους ευθυνών. Γιατί για να προχωρήσουμε, για να αρχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, θα πρέπει να έχουμε πείγνωση του πόσα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ήδη. Έγιναν πολλά, δηλαδή έχει αναγνωριστεί ότι είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της ε, βίας των γυναικών. Αυτό έδωσε όθηση παροκίνησε, παρότρινε πολλές χώρε ε, να κάνουν τι πρωτοβουλίε σαν αυτέ που ακούσαμε, σαν αυτές που υπάρχουν σε άλλες χώρε, ε, Χρειαζόμαστε νομοθεσία, χρειαζόμαστε προληπτικέ πολιτικές, ε, πολιτικές λοιπόν, πρόληψη αλλά και παροχής βοήθειας στα θύματα. Χρειαζόμαστε όμως και εκπαιδευτικέ πολιτικές για να αλλάξει η κοινωνία αυτή που γι' αυτό χρειάζεται όθηση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό οι εμπειρίες σαν τη σημερινή να ληφθούν υπόψη, όπου έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρών. Απευθύνω έκκληση στην Επίτροπο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν από εδώ να δρομολογήσουν πρωτοβουλίες Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα νομικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε στον αγώνα μας ε, για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Και σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Η Ρομπέρτα Μέτσολα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπω και οι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλου του προσκεκλημένους για τι πολύ σημαντικέ πληροφορίε που ακούσαμε. Η βία κατά των γυναικών ε, πολύ συχνά αποσιωπάται, πολύ συχνά την ανεχόμαστε και χρειάζεται λοιπόν μια ε, συνοχή, ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία. Η ομάδα του ΕΛΚ λοιπόν εξακολουθεί να παροτρύνει όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης. Τώρα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο και να πω ότι είναι ευθύνη μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να, για να τιμωρήσουμε την ατιμορρησία και τους ε, δράστες της έμφυλης βίας. Νομίζω πως υπάρχει κοινή συνένεση στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω όμως και μία έτσι πιο πρακτική ερώτηση προς την ε, κυρία Χάιμερ και την κυρία Έκστρομ. Αναφερθήκατε στον πολύ μεγάλο αριθμό ε, ατόμων που καλούν αυτό τον αριθμό εκτακτής ανάγκης. Εγώ θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το προφίλ αυτών των γυναικών που ε, καλούν, που ε, συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Θα ήθελα να μάθω για την εθνικότητά τους, για το μορφωτικό επίπεδο. Μας είπατε ότι αυξήθηκαν οι κλήσεις από μη Σουηδούς υπηκόους Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω τις ε, δικές σας ε, εμπειρίες. Τι σας λένε αυτές οι γυναίκες όταν καλούν αυτόν τον αριθμό. Ε, και μετά, όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, πολύ συχνά μας έρχονται στο μυαλό οι σύζυγοι που βιοπραγούν στις γυναίκες τους. Υπάρχουν όμως και οι γονείς, οι πατέρες που χτυπούν τα παιδιά τους, κορίτσια και γόρια. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, ε, έχετε συναντήσει ποτέ περιπτώσεις που παίρνουν κορίτσια τηλέφωνο και μιλάνε ε, για το ότι όχι μόνο οι ίδιες αλλά και τα αδέρφια τους έχουν πέσει θύματα βίας. Υπάρχουν... Ε, Υπάρχουν τμήματα ή πάλι που ασχολούνται με τα αγόρια ή μόνο με τα κορίτσια ασχολείστε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέντια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και από μένα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους για αυτά που ακούσαμε. Χρειάζεται συνεργασία όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνικό επίπεδο, διασυνοριακό έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα όμως να τονίσω τρία πράγματα από αυτά που άκουσα σήμερα. Καταρχάς, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο ένα ε, ε, ρηξικέλευτο έγγραφο, αλλά είναι καινοτόμο ακριβώς γιατί δείχνει ότι η πολυμερή συνεργασία έχει αποτέλεσμα και μπορεί να επιφέρει την πρόοδο σε πολλούς τομείς της πολιτικής. Ιδιαίτερα μάλιστα, μάλιστα σε εποχές εθνικής πόλωσης νομίζω πως μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μαζί. Αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως βλέπουμε ότι η ε, πολυμερή συνεργασία είναι κλειδί. Μετά το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι οι εκστρατείε ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάνουν τα όρατα θέματα ορατά και δείχνουν ότι δεν σταματάμε σε εκδηλώσεις, συζητήσεις, έτσι, φωτογραφίσεις στις 25 Νοεμβρίου, ας πούμε, την επέτειο, αλλά ε, αναλαμβάνουμε και δράση νομική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ε, έχει η κοινωνία. Και νομίζω πως η προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο ε, για μα στην Επιτροπή Γυναικών, αλλά για όλου. Και εμεί τη Επιτροπή Γυναικών πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να πιέσουμε για οδηγία κατά τη έμφυλη βία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, νομίζω πω πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία έχουμε ένα πρόεδρο που λέει ότι εντάξει, αν πιάνει μια γυναίκα από τα γενετικά τη όργανα δεν τρέχει και τίποτα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι μόλις εγκρίθηκε ένας νόμος από τη Δούμα που αποποινικοποιεί εν μέρη την ενδοοικογενειακή τη δουμα που αποποινικοποιει εν μερει την ενδοοικογενειακη βια είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συζητηθεί το θέμα, να, γίνει, να γίνουν δράσεις γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ της ταχύτατης προσχώρηση της σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά και δεν ε, στρουθοκαμιλίζει. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή γίνεται. Λες και είμαστε το πρώτο κοινοβούλιο που θα κυρώσουμε αυτή τη σύμβαση παγκοσμίω. Ενώ ξέρουμε ότι είναι πολλά τα κράτη-μέλη που έχουν ε, προσχωρήσει. Περίπου τα μισά έχουν κυρώσει. Η Πολωνία, η Λιθουανία, η Γαλλία έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι προφανές η καταπολέμηση της ομοφικογενειακής βίας. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ποια είναι η συλλογιστική πίσω από το να κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύμβαση αυτή η νομοθεσία ε, και γενικώ το δίκαιο προβλέπει ότι δύο φορεί δεν μπορούν να έχουν ταυτόχρονα τι ίδιε αρμοδιότητε. Ω Ένωση Κρατών, αν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τι αρμοδιότητε, αλλάζουν τα πράγματα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει λοιπόν να υποστηρίξει τα κρατημέλη στην καταπολέμηση τη ενδοικογενειακή βία και να εφαρμόσει κάποια μέτρα της σύμβασης, όπως, χάρη, όπως λόγω χάρη τους πολιτιστικούς, τα πολιτιστικά αίτια που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ των γεννασιωργών ε, αιτίων, ε, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν κοιτάζουμε τα πολιτιστικά ε, αίτια λόγου χάρη ή δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στην όλη συζήτηση η πορνογραφία. Ε, η πορνογραφία ε, πραγματικά επιτρέπει και καλλιεργεί πολλέ μορφέ βία κατά των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, όμω ποιο είναι ο σκοπό τη κύρωση τη ε, σύμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι και πάλι ε, δεν είναι καλή ιδέα να ε, έχουμε ακριβώ τι ίδιε αρμοδιότητε με τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, θα είναι σε πλήρη αντίθεση με το κράτο δικαίου που πρέπει να σεβαστούμε. Δεν μπορεί λοιπόν τα ίδια καθήκοντα να παραλαμβάνουν δύο φορέ ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμε. Να ευχαριστήσω και εγώ τις προστακλημένες μας για την τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη επισκόπηση και παρουσιάση που μας έκανα για να καταλάβουμε την πραγματική σημασία του να κυρώσει η Ένωση και όχι απλώς τα κρατη στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ελπίζω ότι αυτό θα σημαίνει πραγματική δράση την διαδικασία αυτή εκμάθησε στην πραγματικότητα που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για να καταφέρουν να καταπολεμήσουν την ενδοκογενειακή βία. Να ρωτήσω τις προσκεκλημένες μας, εάν μπόρεσαν στις μελέτες τους, στην πρακτική τους εμπειρία, να εντοπίσουν τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης πώς επηρέασε κάτι κράτη-μέλη όλος ιδιαίτερος. Τι συνέπειες είχε τη σχέση με την ενδοκογενειακή βία και το τεράστιο άγχος και την τεράστια δυσφορία που έχει προκαλέσει στην κοινωνία. Το βλέπω να συμβαίνει στη χώρα μου. Μια από τις χώρες που έχει χτυπηθεί πολύ σκληρά από την οικονομική κρίση τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόστηκαν, ο αντίκτυπος που υπήρχε στις διάφορες οικογένειες, με τεράστιες μορφές βίας να αναζωπυρώνονται και βεβαίως η βία στις οικογένειες, κυρίως αστέφεται κατά των γυναικών και των παιδιών. Επίσης με κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών στα πλαίσια της αντικογενειακής βίας. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με κάτι που ήδη υπόθηκε. Οι επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης της Ντούμα, η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ποινικοποιήσει στην ουσία, να νομιμοποιήσει την ενδοκοκενιακή βία. Έχετε σκεφτεί τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η απόφαση, όχι μόνο στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της ευρύτερης αυτής γεωγραφικής περιοχής. Μπορεί να αισθανθούν ε, την άνεση να, να, να κάνουν κάτι εξίσου απολύτιστο. Ευχαριστούμε κυρία Γουόρντ. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να πω και εγώ ότι είναι πραγματικά πολύ ευχαριστώ να ακούει κανείς τις παρουσιάσεις τόσο έγκριτων εμπειροχονομόνων και ειδικών με βέλτιστες πρακτικές που μας στάνουν λόγω χάρη από τη Σουηδία. Ταξιδεύω και συναντώ γυναίκες από όλα τα κράτη-μέλη. Και ήθελα εδώ να μιλήσω με τη δική τους φωνή, διότι πραγματικά ε, καλούν ε, απεγνωσμένα για δράση αυτά τα κράτη-μέλη. Όταν τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται να κυρώσουν μια τέτοια σύμβαση ή να την κυρώσουν χωρίς να την εφαρμόσουν, οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να στραφούν σε έναν άλλο φορέα που θα ε, ψώσει το ανάστημά του, ζητώντας τα, γυναί... τα δικαιώματα, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι δικαιώματα ανθρώπινα. Μια από τις ε, γνωστές μου ακτιβίστρια σε μια από τις χώρες για τα γυναικεία δικαιώματα, δεν θα πω σε ποια χώρα, είπε η χώρα μου δεν θα κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, διότι κοστίζει. Και η απάντησή μου είναι, το κόστος είναι οι ζωές των γυναικών. Έχουμε συζητήσει εδώ για το οικονομικό κόστος κάποιες φορές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους, λόγω της βίας που ασκείται εναντίον τους. Αυτό θα πρέπει να το καταγράψουμε ως δεδομένο στη σημερινή συζήτηση, στη σημερινή κουβέντα. Έχουμε καθήκον ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα, ως ε, μέλη Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου να προασπιστούμε και να προστατεύσουμε τις αδερφές μας που κινδυνεύουν. Πολλές επιθετικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα κράτη-μέλη που ουσιαστικά ε, διαλύουν τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν αρκεί να ακυρώσουμε. Πρέπει και να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση με διάφορες διαδικασίες μετά την προσχώρηση. Θέλω λοιπόν να σταθώ λίγο και στα μέτρα λιτότητας, τα έθιξε και η Άννα. Τα μέτρα λιτότητας συνεισέφεραν ιδιαίτερο στην, ε, στην ε, ένταση, την μεγαλύτερη εξάπλωση της βίας εντός των οικογενειών, αλλά υπάρχουν και περισσότερες ε, επιπτώσεις λόγω των προσφύγων, των μεταναστιδών, της μικρότερης διάθεσης υπηρεσιών προς τις γυναίκες λόγω οικονομικής πίεσης. Αυτό συνέβη και στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οικονομικές πολιτικές επηρεάζουν την κατάσταση των γυναικών. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι γίνεται και με την ε, ε, εφαρμογή των προτύπων που έχουν να κάνουν με τη στάση των μαρτύρων όσων είναι μάρτυρες μορφές βίας κατά των γυναικών και δεν καταγγέλουν, δεν τα εντοπίζουν. Επίσης η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τις σεξουαλικές ε, σχέσεις και την ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ανδρών και γυναικών. Πρέπει να μιλήσουμε για όλες τις μορφές βίας που γνωρίζουν οι γυναίκες. Ευχαριστούμε η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την ε, βία κατά των γυναικών. Πρέπει και να προλαμβάνετε και να καταπολεμάτε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις προσκεκλημένες μας σήμερα το απόγευμα και θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα οι γυναίκε με ειδικέ ανάγκε έχουν πρόσβαση στι διάφορε υπηρεσίε που διατίθενται. Λόγου χάρη, φανταστείτε μια γυναίκα που έχει προβλήματα ακοή και έχει υποστεί τέτοιου είδου βία. Δεν μπορεί να πάρει την γραμμή αυτή για τα θύματα. Την ειδική τηλεφωνική γραμμή. Τι θα κάνει. Εγώ επίσης είμαι κοφάλαλη. Αυτό είναι ένα επιπλέον εμπόδιο που κάνει τη ζωή ιδιαίτερα δύσκολη. Και όπως και η σεξουαλική βία υπάρχει και το θέμα των ε, εστιών. Εκεί που μπορούν να απευθυνθούν αυτοί που έχουν ειδικέ ανάγκε λόγου χάρη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για τι γυναίκε γενικώ, αλλά οι γυναίκε με αναπηρίε έχουν να υποστούν ακόμη μεγαλύτερη διακριτική μεταχείριση. Και αν μιλάμε για γυναίκε πρόσφυγες έχουν τις απαραίτητε πληροφορίε για να ξέρουν πού να απευθυνθούν, για τις φροντίζεται για τις γυναίκες πρόσφυγες, είναι μια ειδική κατηγορία και αυτές. Στην Σουηδία, στις Βρυξέλλες, αλλού. Οπουδήποτε. Γνωρίζουν οι γυναίκες τι υπηρεσίες προσφέρονται και τέλος για το θέμα της κύρωσης και της προσχώρησης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη. Ποια είναι η προστεθέμενη αξία της ε, προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βεβαία ότι υπάρχει αυτή, αλλά μπορείτε να μας την εξηγήσετε στα ράτα. Ε, ποια είναι η διαφορά. Βλέπουμε ότι 14 κάτι μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση και τα υπόλοιπα όχι. Ε, άρα ξαφνικά μου γεννάται η απορία γιατί. Γιατί δεν την έχουν κυρώσει. Διότι είναι σαφές ότι η κύρωση της Κωνσταντινούπολης είναι σημαντική. στην ε, Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ας πούμε, ε, είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες χώρες όπου είναι εντονότερη η βία κατά των γυναικών. Δεν είναι απλώς δηλαδή το θέμα η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και της ανταλλαγής απόψεων. Θα σας ήμουν ευγνώμων να μας δώσω δίνατε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε κυρία Χάνιμπολ. Uh, uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τις συζητητές και όλους τους ε, ομιλητές. Όπως γνωρίζουμε, η έμφυλη βία, βία κατά των γυναικών, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε τι έκταση έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω πως ε, οι δύο επιτροπές μας πράγματι κάνουν βήματα προς την προσχώρηση στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν μένουν εκεί. Ασχολούνται γενικά με την αντιμετώπιση της έμφυλη βία. Μάλιστα, εγώ να σας πω ότι προσωπικά ντρέπομαι που μόνο 14 κράτη-μέλη έχουν επιχειρώσει την σύμβαση. Το, η δικιά μου χώρα ανήκει σε αυτές. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει τι δουλειά πρέπει εμείς να κάνουμε και 14 κράτη-μέλη τι σημαίνει, το 50%. Μόνο τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Το πρόβλημα αυτό είναι λοιπόν. Τα άλλα 14 τι κάνουν, γιατί καθυστερούν. Και θεωρώ πως ε, η δική μας προσπιθέμενη αξία ε, είναι η άσκηση πίεσης στα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση να το πράξουν. Να τους πούμε δηλαδή ότι κοίταξε, εμείς το κάναμε. Εσείς πότε αυτή νομίζω είναι η δική μας προστιθέμενη αξία. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης, ε, τη οποία την 60η επέτειο μόλις γιορτάσαμε κιόλας. Η επετειο μόλι γιορτασαμε κιόλα. έχει ήδη δηλαδή κάνει την αρχή και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι και να παραδεχτούμε ότι από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει όσο θα έπρεπε. Νομίζω μια προηγούμενη ομιλήτρια αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ο μισογυνισμός και το μίσος ξεκάθαρα κατά των γυναικών γίνεται όλο ένα και πιο φθαλμοφανές σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης. Δεν θα πω προφανές, οφθαλμοφανές. Και η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται. Το καλό όμως είναι ότι αρχίζουμε να συζητάμε γι' αυτό ανοιχτά και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ και πέρα από την επικύρωση της Συμβάσης Κωνσταντινούπολης. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, μία οδηγία κατά της έμφυλης βίας, διότι πιστεύω πως έχουμε εδώ την ευκαιρία να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και δεν πρέπει να, ε, να μην ε, πάρουμε αυτή την ευκαιρία στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινής, ε, αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Η συνάδελφος κυρία Χάνιμπολ αναφέρθηκε ήδη σε αυτό, ότι δηλαδή Πέρασαν πολλά χρόνια, δεκαετίες αιώνες μέχρι να παραδεχτούμε το φαινόμενο της ε, βίας κατά των γυναικών. Μέχρι τώρα σιωπούσαμε και οι γυναίκες πολύ συχνά δεν μπορούσαν να βρουν κανένα να τι βοηθήσει. Δεν είχαν στήριξη από τις οικογένειές τους και αναγκάζονταν να ε, πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν είχαν εναλλακτική λύση. Πράγματι λοιπόν άλλαξαν κάποια πράγματα, ωστόσο συνεχίζουμε να ε, βιώνουμε θέματα βίας ε, κατά των γυναικών. Είναι καθημερινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βία κατά των γυναικών και τα μέσα ενημέρωσης γράφουν γι' αυτό, όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και βίας ε, στον στενό κύκλο των γυναικών, από τους γείτονες, τους, το φιλικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δώσουμε το καλό παράδειγμα και βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά της έμφυλης βίας ολοένα και μειώνεται. Γίνονται περικοπές εξαιτία της κρίσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να λαμβάνουν να παρκεί χρηματοδότηση αυτά τα προγράμματα. Θεωρώ πως είναι αναγκαίο να τονίζουμε, να αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα ε, για την βία, όχι μόνο σε τρίτες χώρες που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλο τρόπο ζωής κτλ, αλλά και εδώ, στο δικό μας το σπίτι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η κυρία Χάνιμπολ, δεν έχουν επικυρώσει, δεν έχουν υπογράψει μάλλον ε, όλα τα κράτη-μέλη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μόνο τα μισά. Γι' αυτό ε, λοιπόν ε, είναι σημαντικό. Και επίσης τα κράτη που την έχουν υπογράψει δεν, ε, προσπα... δεν την έχουν επικυρώσει ακόμα, δεν βιάζονται. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα αυτό πιο προσεκτικά. Τώρα, οι ποινέ. Οι ποινέ είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί. Νομίζω πω ο ορισμό καταρχά ε, τη είναι προβληματική. Υπάρχει και μία φράση, εγκλήματα τιμή, φόνη τιμή. Ε, νομίζω πω αυτό είναι από μόνο το προβληματικό. Δεν υπάρχει καμία τιμή στο να σκοτώνει μία γυναίκα. Είναι σκέτο φόνος. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό είναι συνδεδεμένο με την κουλτούρα, με τις πεπιθήσεις, με οτιδήποτε. Είναι φόνος απλά τελεία και παύλα. Πρέπει όμως να, γι, ε, να γίνουν πολλά στις ίδιες μας τις χώρες, ενημέρωση των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή την πτυχή της επικύρωσης της συνθήκης ως Κατινούπολης να την χρησιμοποιήσουμε, την ενημέρωση δηλαδή, την ευαισθητοποίηση έτσι ώστε να γίνει πρόοδος και να βγουν οι γυναίκες από αυτό τον εφιάλτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο τους προσκεκλημένους μας και θα αρχίσουμε με την κυρία Γκαφαρόβα. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες μας τις, όλες τις βουλευτές και τους βουλευτές. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα και να ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Κάποιος ανέφερε εδώ ότι το θέμα της κύρωσης είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Όντω, τα περισσότερα διεθνή κύματα, η ισότητα των φύλων και οι θεμελιώδει ελευθερίε θεωρούνται τα θεμέλια της κοινωνίας. Το θέμα με την ισότητα των φύλων είναι ένας δείκτης για το πόσο είναι ανεπτυγμένη η δημοκρατία στη μία ή την άλλη χώρα. Υπόθηκε ότι η την αλλη χωρα υποθηκε οτι η συμφωση της Κωνσταντινούπολης έχει κυρωθεί από κάποιες χώρες, ε, έχουν προσχωρήσει. Κάποιοι δεν έχουν προσπογράψει ούτε ε, την έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Εγώ υπό την ιδιότητά μου πρέπει να πω ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και βεβαίω την όλη αυτή συζήτηση πρέπει να ε, έχουμε υπόψη ότι Προφανώς πρέπει να δώσουμε αγώνα για το θέμα αυτό. Οι γυναίκες ε, πρέπει να έχουν ως το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία στο διεθνές δίκαιο. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές φορές αυτά τα δεδηλωμένα ίσα δικαιώματα δεν γίνονται πραγματικότητα, διότι ακριβώ δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Πρέπει λοιπόν τα ίσα δικαιώματα να είναι πραγματικότητα και στην νομοθεσία μας και στις κοινωνίες μας. Ευχαριστούμε η κυρία Μουαρό Μπρό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό και το υπογράμμισαν πολλοί ομιλητές. Πολύ περισσότερες χώρες να προσχωρήσουν στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης και όσες έχουν προσχωρήσει και υπογράψει να την επικυρώσουν βέβαια. αν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. φυσικά αυτό θα δώσει παρότρινση και στα άλλα κράτη. Αυτό το προκαταρκτικό σχόλιο. Μίλησαν κάποιοι για τη χρηματοοικονομική κρίση, τα πρόσεξα αυτά τα σχόλια, σε σχέση και με τις γυναίκες, ε, τις μετανάστριες γυναίκες. Και πράγματι, Κάθε φορά που οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες βέβαια βρίσκονται σε μια επισφαλή κατάσταση και ιδίως βέβαια εδώ οι γυναίκες, αυτό επιδεινώνει τα φαινόμενα βίας. Άρα εδώ τη θέμα θα αντιμέτωπε με το φαινόμενο οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν περισσότερα ε, κρούσματα βίας επειδή είναι πιο ευάλωτες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να κατασταθεί αυτός ο παύλος κύκλος. Περισσότερες οικονομικές δυσχέρειες να οδηγούν σε περισσότερη βία, επομένως δυστυχώς και σε μεγαλύτερη επισφάλεια. Αν σε αυτό το, το τέλος της αλυσίδας αυτής δεν υπάρχει μία προστασία, μία υποστήριξη για τις γυναίκες, δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας. Ε, πολύ σωστά υπογραμμίστηκε ότι οι βολονταριστικές πολιτικές για την υποστήριξη των ε, γυναικών που είναι θύματα βίας, δηλαδή καλύτερη συνθήκες ε, φιλοξενίας ε, διαμονής, βοήθεια καλύτερη για να μπορέσουν να φύγουν από την αιστεία τους, εφόσον εκεί υφίστανται την οικογενειακή βία κτλ. Πρόκειται για δαπανηρά μέτρα. Ισχύει αυτό. Όμως, κάποιος είπε ότι οι γυναίκες που είναι θύμα βίας, που μπορεί να χτυπηθούν μέχρι θανάτου ή να υποστούν ψυχολογική βία και όχι μόνο σωματική. Αυτό συνιστά τεράστιο κόστος για την κοινωνία και πρέπει να το έχουμε υπόψη και να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι για το ότι τα προβλήματα αυτά μετακυλίονται ε, στον τομέα της υγείας και σε πολλά άλλα επίπεδα. Και στα παιδιά βέβαια. Οπότε Πρόκειται όχι μόνο για το μέλλον των γυναικών, αλλά και για το μέλλον όλων ανδρών και γυναικών, τα παιδιά, για τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν κάθε κράτος μέλος ε, να βοηθήσει και στη χρηματοδότηση και στα απαραίτητα μέτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Καθηγήτρια Γκάι, Χάιμερ. Ευχαριστώ σε ό,τι είπατε ε, για τη τηλεφωνική γραμμή από τη ηλικία των 16 ε, κορίτσια και όχι άνδρες και ούτε και παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γραμμή. Και φυσικά υπάρχει ανωνυμία, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί ε, το κορίτσι αυτό να μιλήσει για πρώτη φορά για αυτή τη μορφή βίας, άρα θα πρέπει να είναι ανώνυμο το τηλεφώνημα. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα τιμής και τη βία, οι περισσότεροι που τηλεφωνούν στη γραμμή βοήθειας είναι Σουηδέζες γυναίκες ε, από τη Σουηδία. Ε, αναφέρει και τα θέματα της αναπηρίας. Οι γυναίκες που έχουν και κάποια αναπηρία σίγουρα είναι πιο περιθωριοποιημένες σε σχέση με τις Και είναι γεγονός ότι οι δράστες, ε, οι άνδρες, μπορεί να ανήκουν στην οικογένεια, αλλά να είναι και ίσως και φροντιστές της γυναίκας αυτής. Ε, άρα να και μια ακόμη κατηγορία που πρέπει να έχουμε υπόψη. Και έχουμε κάνει έρευνες και φαίνεται ότι ιδίω οι πιο ηλικιωμένε γυναίκες ε, είναι ευάλωτη ομάδα πλέον. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε στη συζήτηση, μιλάμε και για ένα έγκλημα εμπιστοσύνης, διότι η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν βοήθεια ε, και μετά ζητάμε από αυτές τις γυναίκες να έρθουν και να μας πούν ε, τι τους συμβαίνει. Πρέπει να προσεγγίσουμε τις γυναίκες, να δούμε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο, ότι οι γυναίκες ε, πρέπει να πιστούν ότι τους λαμβάνουν, τις λαμβάνουν σοβαρή υπόψη. Θα πρέπει να υπάρχουν εμπειρογνώμονες και στην αστυνομία και στο δικαστικό σώμα. Εφόσον η βία είναι έγκλημα, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση, να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα θύματα της βίας για να τα βοηθήσω. Και η συζήτηση σήμερα δείχνει τη μεγάλη σημασία του θέματο. Πεθαίνουν γυναίκες στην Ευρώπη και στη Σουηδία και στη Φινλανδία και στη Δανία. Έχουμε δει πολύ ψηλά νούμερα τα κρούσματα και μιλάμε για χώρες με τα μεγαλύτερα ε, ποσοστά τα υψηλότερα ποσοστά ισότητα. Άρα χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση για να έχουμε πρόσβαση στου ευάλωτου αλλά θα πρέπει να πιστεύουμε ε, σε αυτό που κάνουμε και να πιστεύουμε στη Σύμβαση Κωνσταντίνου Γιατί αυτό δεν φέρνει να αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Μιγγέλ Σιέρα. Μιλήσαμε πριν για γυναίκες με αναπηρία. Δεν υπάρχουν ακόμη δομές που να μπορούν να φιλοξενήσουν τις γυναίκες αυτές με παρκή, με, με το κατάλληλο τρόπο. Υπάρχει όμως ε, και το άλλο θέμα που το αναφέραμε, ότι μόλις τώρα άρχισαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα για τις γυναίκες ε, που είναι στο δρόμο, τις άστεγες, για τις γυναίκες με αναπηρία, για τις μετανάστρες, τις πρόσφυγες, για ε, τα κορίτσια που μπορεί να είναι θύμα μπορεί να ε, έχουν αναγκαστεί να παντρευτούν κτλ. κτλ. Τώρα αρχίζουμε να το πιάνουμε το θέμα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να επιστήσουμε την προσοχή στην πραγματικότητα αυτή, που δεν θέλουμε να τη βλέπουμε. Δεν θέλουμε να τη βλέπουμε και δεν θέλουμε να τη μετρήσουμε. Το θέμα το... Ε, περιορίζουμε στο να πούμε αν είναι εθνικό θέμα και τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν μεγάλες χώρες που ουσιαστικά υπονομεύουν τις προσπάθειες για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Σίγουρα και είναι κατεπήγον και πρέπει να... Φυσικά και χρειάζεται ένα πολύ στέρεο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ε, μορφών βίας κατά γυναικών και παιδιών. Και φυσικά η επικύρωση, η προσχώρηση είναι ένα πρωτό σημαντικό βήμα. Ευχαριστώ. Thank you. And now, uh, Mrs. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Ρεβόνταλόν Μπονφουά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά να πω ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να έχουμε τις πληροφορίες, ε, τις ειδικέ αυτές όσων εργάζονται επιτόπου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως είπατε και εγώ είμαι βεβαία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρωπαϊκός ε, θεσμός πρέπει να κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι κάτι το αξιοπερίεργο και ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Για το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κυρώσει και ε, προσχωρήσει στην σύμβαση του ΙΕ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις γυναίκες. Τον μισό πληθυσμό της Ένωσης, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα αναμιμότητα ούτε θεμητού, ώστε να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και λαμβάνοντα υπόψη την τόσο μεγάλη ανισότητα των ε, γυναικών ασχέτα, ασχέτως του τόπου διαμονή διαμονής τους. Όπω είπε και η κυρία Μάνο, ε, γιορτάσαμε τα 60 χρόνια από τη συνθήκη τη Ρώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει περισσότερο του Ευρωπαίου πολίτε και τι Ευρωπαίε πολίτε. Είναι άκρο σημαντικό. Η κύρωση τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη είναι ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο, που είναι επίση αναγκαίο, θα είναι μια οδηγία, ώστε να έχουμε και το νομοθετικό πλαίσιο για να είμαστε βέβαιοι ότι οι γυναίκε έχουν τα ίδια δικαιώματα. Σα ευχαριστώ και πάλι. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μα για την έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους και τα μέλη των δύο επιτροπών για την ενεργό τους δράση, για το ότι ήρθαν εδώ, εξέφρασαν τις απόψεις τους για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. με ενημέρωσαν μόλις ότι μάλλον θα καταφέρει να έρθει η κυρία Κορατσαμπίλ. Να επενθυμίσω όμως σε όλου ότι αυτή η κοινή ακρόαση των Επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Γυναικών θα έχει και συνέχεια, η οποία θα λάβει χώρα στις 12 Απριλίου. Τώρα, ε, καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών για την έκθεση των δύο συνεισηγητριών είναι 26 Απριλίου. 12 το μεσημέρι, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 12 Ιουνίου. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών ότι σε ένα-δύο λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της δικής μας Επιτροπής. We will continue uh, our hearing <laughs> for uh, two or three minutes. Θα συνεχίσουμε λοιπόν για δύο-τρία λεπτά την ακρόαση. Κύριε Κοράτσα Μπίλτ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ που με περιμένατε, γιατί ήθελα πραγματικά να έρθω σήμερα, αλλά κόλλησα στο αεροδρόμιο τη Στοκχόλμη. Η πτήση μου είχε τεράστια καθυστέρηση. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σίγουρα είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα σα ακούσω αργότερα. Θα ήθελα Πάντως να πω ότι εξακολουθούμε να είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για την πολιτική της μηδενικής ανοχής ε, κατά της ε, έμφυλης βία, τη βία, της βίας από άνδρες ε, σε γυναίκες. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους κοιόντες εισηγητές. Μόλις παρουσιάσαμε το σχέδιο έκθεσης και νομίζω πως ήταν και πολύ επίκαιρη η ακρόαση σήμερα. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ε, Σίγουρα αναφερθήκατε στα ουσιώδη. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε με τις εκκρεμότητες και ο ορισμός του φύλου είναι από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε όπως τώρα. Χρειάζεται να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, εφαρμόσουν 100% απόλυτα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να την επικυρώσουν αν δεν το έχουν κάνει, να προσχωρήσουμε με ε, χρησιμοποιώντας ε, το μεγαλύτερο δυνατό εύρος. Εάν συνεχίζουμε αυτή την ε, πρακτική των εξαιρέσεων, των δισταγμών, των παρερμηνιών, τότε δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τι σημαίνει η έμφυλη βία, το φύλλο, βία κατά των γυναικών. Αυτό ζητά και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, που ε, είναι και κτήμα του κιόλας η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλοσοφίες. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γίνει έκκληση, έχει γίνει έκκληση και προς τα κράτη-μέλη μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης να ε, ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος για να δούμε τα προβλήματα και να βρούμε τις λύσεις. Δεν έχει να κάνει ούτε με χριστιανικές αξίες, ε, ούτε με τίποτα τέτοιο. Γυναίκες, κορίτσια, ε, υφίστανται βία, βιάζονται. Η έμφυλη βία δεν είναι ε, κάτι που συζητάτε και κλεισμένον των θυρών. Η έμφυλη βία είναι έγκλημα, ποινικό αδίκημα και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πως χαίρομαι πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από την κοινωνία των πολιτών και να συγχαρώ και τις συναδέλφους από τη Σουηδία γιατί η δράση είναι υποδειγματική ε, του κέντρου αυτού. Ενημερώνει, προστατεύει, καταρτίζει, εκπαιδεύει. Κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ανεξάρτητα από σε, το σε ποια πολιτική ομάδα ανήκουμε, για να ακουστεί η φωνή μας στα κράτη-μέλη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο θα σταματήσω, ωστόσο με μεγάλη μου χαρά να συζητήσω μερό με όποιον το επιθυμεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κορατσαμπίλτ. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών.